στήσιμο των αγώνων και η διαφθορά στον αθλητισμό. Έχει το λόγο η κυρία Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το στήσιμο των αγώνων και η διαφθορά είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρωπαϊκός αθλητισμός. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τις αρχές του αθλητισμού να το αντιμετωπίσουν. Οπωσδήποτε γνωρίζω την εμπλοκή των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος στο πιο πρόσφατο σκάνδαλο που επηρεάζει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίε μου έχουν έρθει σε επαφή, με την Ευρωπόλ για να συζητήσουν την υπόθεση και καλωσορίζω την δράση της Europol μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τώρα την ε, σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το στήσιμο αθλητικών γεγονότων, η Κομισιόν το 2012 υιοθέτησε μία σύσταση προς το Συμβούλιο. Η σύσταση αυτή ζητάει από τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις και αναμένουμε το Συμβούλιο να υιοθετήσει τη διαπραγματευτική του εντολή προσεχώς. Θεωρώ πως η ε, σύμβαση όταν υιοθετηθεί θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για την αποφασιστικότητα της Ευρώπης για να διατηρήσει την αγκαιριότητα του αθλητισμού. Επίσης η σύμβαση θα πρέπει να είναι ανοιχτή προς υπογραφή και από μη ευρωπαϊκές χώρες για να δούμε έτσι και την παγκόσμια διάσταση του προβλήματος. Για να έχουμε μια συνολική προσέγγιση όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν συνεργάζονται τώρα στενά για να διασφαλίσουν την ε, συμβατότητα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο πλαίσιο, στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εσωτερική αγορά. Όπως δείχνει και η εμπλοκή της Ευρωπόλ, οι αρχές επιβολής του νόμου και η συνεργασία του στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχει κέρια σημασία για να καταπολεμηθεί αυτή η απειλή. Οι πρόσφατες αυτές περιπτώσεις της σήματος αγώνων θα απαιτήσουν στενή συνεργασία μεταξύ δικαστικών αρχών ε, και στην έρευνα και στην δίωξη. Οι αρμόδιες αρχές θα μπορέσουν να βασιστούν στο Eurojust για την πρακτική ε, συνεργασία και τις διασυνοριακές διώξεις. Αλλά και θα μπορέσουν να βασιστούν σε μια σειρά μέσων που έχουν υιοθετηθεί στον τομέα της ε, δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Όμως, βεβαίω όλα αυτά είναι μία πτυχή της λύσης. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, η καταπολέμηση του στισίματος των αγώνων πρέπει να περιλαμβάνει και προληπτικά μέτρα. Με χαρά μπορώ να σας ενημερώσω πως ε, Σύμφωνα με τι προπαρασκευαστικέ ενέργειες του 2012 για τον αθλητισμό, η Κομισιόν έχει επιλέξει πέντε έργα στον τομέα του στισήματο των αγώνων. Τα έργα αυτά θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση των αρμοδίων και στον τομέα του αθλητισμού και στην κοινή γνώμη. Ε, Ξεκινήσαμε στις αρχές του έτους να εργαζόμαστε πάνω στο θέμα και αναμένουμε αποτελέσματα το πρώτο εξάμεινο του 2014. Οι συντονιστές των έργων αυτών συνεργάζονται για να έχουμε συνέργειες και κοινέ στρατηγικές. Τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να διαδώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να ενισχύσουμε τα δίκτυα. Θα ήθελα επίση να προσθέσω πω συνεργάζομαι στενά με τον συναδελφό μου, τον κύριο Μπαρνιέ, για να δούμε το ζήτημα του στισίματος από την πλευρά των ε, στοιχημάτων. Στις 23 Νοεμβρίου του 2012 η Κομισιόν υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης ε, για τον ε, τζόγο στο διαδίκτυο που περιείχε και ένα κεφάλαιο για την ακαιρεότητα στον αθλητισμό. Αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν μεταξύ άλλων είναι μια σύσταση που θα υιοθετηθεί το 2014. Η σύσταση αυτή θα ενθαρρύνει μια πιο αποτελεσματική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην πρόληψη και καταπολέμηση του στισίματος από την πλευρά του στοιχήματος. Οπότε καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία να συνεισφέρουν στην διαμόρφωσή της. Επίσης θα έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες όπως ε, μελέτες, εργαστήρια, συναντήσεις ειδικών για την συγκέντρωση στοιχείων και την ε, καλύτερη σύνταξη της σύστασης. Τέλος, στις 5 Φεβρουαρίου τρέχοντος ε, προτείναμε την χρήση της ε, οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρωμίκου χρήματος, καθώς ε, ο τομέας ε, του στοιχήματος είναι ευάλωτο στο ξέπλυμα βρωμικού χρήματος και προτείναμε πέρα από τα καζίνο να καλυφθεί όλος ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών δεδομένης εξέλιξη του ξεπλήματο χρήματο είναι σημαντικό το ευρωπαϊκό πλαίσιο να μπορεί να ανταποκριθεί με τρόπο εύρωστο και ευέλικτο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Περνάμε στου ομιλητές εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων για την ε, ομάδα του ΕΡΤ για δύο λεπτά κύριο Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι και θέλω να ευχαριστήσω και την ε, Πέτρα Κάμερεβερτ και τον κύριο Λόκεγκαρντ για αυτή την ε, πρωτοβουλία στα Ολλανδικά τώρα. Ε, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι βεβαίως καταδεικνύει πως η... το στήσιμο αυτό αποτελεί μια μεγάλη απειλή για τον αθλητισμό στην Ευρώπη και χρειάζεται μια προσέγγιση η οποία θα είναι και διεθνής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρξει μια άμεση και δομημένη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αυτών που κάνουν τα στοιχήματα αφενός των ε, ομοσπονδιών, των αθλημάτων και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για να είναι αυτόματη, όπως είπα, η ανταλλαγή των δεδομένων για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δεύτερον, με το ψήφισμα αυτό, κυρία Επίτροπε, ζητάμε συγκεκριμένα μια νομοθετική πρωτοβουλία της Κομισιόν για να καταπολεμηθεί η απάτη στον αθλητισμό ε, πανευρωπαϊκά και ξέρετε πως σήμερα εκμεταλλεύεται το οργανωμένο έγκλημα την ε, κατάσταση, δηλαδή το ότι έχουμε ένα νομικά κατακαιρματισμένο τοπίο. Οπότε το στίχημα ή απάτη στον αθλητισμό πρέπει να καταπολεμηθεί με συγκεκριμένες και ενιαίες κυρώσεις. Ε, τρίτον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ αυστηρά τα παράνομα site που δεν έχουν άδεια, δεν έχουν καταγραφεί για να μπορούν οι πολίτες που θέλουν να σχηματίσουν να το κάνουν με τρόπο κανονικό. Και τέλος χρειάζεται μια απαγόρευση για το στίχημα των ανηλίκων, η οποία θα είναι πανευρωπαϊκή και θα έχουμε έναν ε, κώδικα συμπεριφοράς για όλους τους συμμετέχοντες ε, όπου θα λένε πως δεν είναι δυνατόν να στοιχηματίζουν οι ανήλικοι. Το σκάνδαλο αυτό με τον τζόγο δείχνει πως ε, δεν επαρκούν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και έχει φτάσει η ώρα να ανεβάσει ταχύτητα η Κομισιόν και οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο θα σας στηρίξει. Αναμένουμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες σας στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Μπέλετ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, μισή λεπτό, η κυρία Κάμερεβέρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, οι έρευνε και οι ανακρίσει έχουν αποκαλύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τουλάχιστον 380 ποδοσφαιριστές έχουν χειραγωγήσει παιχνίδια και αν το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάνω από 700 άτομα και για την Ευρώπη όλοι θεωρούμε ότι είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Δεν μπορούμε να δούμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα πόσο μεγάλη είναι η έκταση αυτού του σκανδάλου. Αυτό είναι ένα πραγματικό ράπισμα στην ιδέα ότι το ποδόσφαιρο και γενικά τα αθλήματα είναι ένας χώρος δίκαιου ανταγωνισμού που προωθεί τις ανθρώπινες αρχές. Η χειραγώγηση και τα παράνομα στοιχήματα καταστρέφουν τελείως αυτή την εικόνα. Θα πρέπει οι οπαδοί να ξέρουν ότι η ομάδα τους αγωνίζεται δίκαια και κερδίζει ή χάνει. Το fair play δεν πρέπει να είναι μονάχα μία δήλωση, μία φράση αλλά και μια πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε πρόληψη, χρειαζόμαστε εποπτεία, αλλά χρειαζόμαστε και κυρώσει. Πρέπει οι Αθλητικέ ενώσει να εφαρμόσουν μια πολιτική μηδενική ανοχή που να βασίζεται σε κοινού κώδικε και τη δημιουργία ενό πλήρου προγράμματο για την πρόληψη τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για ήττα ή νίκη στον αθλητισμό, αλλά και για πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχουν οι δυνατότητε να γίνονται στοιχήματα τα οποία οδηγούν σε χειραγώγηση των αγώνων και θα πρέπει να απαγορευτούν. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο τρόπο να καθορίσουμε τι σημαίνει χειραγώγηση των αγώνων και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κολλάζουν αυτέ τι μορφέ χειραγώγηση των αγώνων. Χρειαζόμαστε και πιο στενή συνεργασία για να υπάρχει καλύτερη δίωξη αυτών των αδικημάτων και θα πρέπει επίση να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και με κανόνε νομοθετικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Επίτροπο για την υποστήριξή της και πιστεύω και ελπίζω ότι το ψήφισμά θα μπορέσει να συμβάλλει στο να γίνουν παρελθόν οι χειραγωγήσει στον αθλητικό τομέα στην Ευρώπη και αλλού. Ευχαριστώ κυρία Κάμερεφετ, λέει ο πρόεδρο. Για δύο λεπτά έχει το λόγο από την φιλελεύθερη ομάδα ο κύριος Λόκεγκάρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ είναι μια θετική ημέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν πρόκειται για τον αγώνα κατά του στισίματος των αγώνων. Αυτά που ακούσαμε από τον, από τον εισηγητή και την Κομισιόν είναι σοφά και εύστοχα και έγκαιρα λόγια. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε όμως πέραν αυτών είναι να προχωρήσουμε και να πάρουμε απτά μέτρα στον αγώνα κατά του στισίματος, όπως είπε και ο εισηγητής, όπως είπε και η Κομισιόν. Αυτό είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου. Είναι μονάχα το ορατό τμήμα μιας μεγάλης μορφής κινδύνου για τον αθλητισμό. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το στήσιμο του αγώνα θα έχουμε τεράστια προβλήματα γιατί πρόκειται για μια πολυπλόκαμη μορφή χειραγώγησης από την Ανατολική Ασία μέχρι τα Βαλκάνια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μορφή οργανωμένου εγκλήματο, το οποίο υποσκάπτει τα θεμέλια του αθλητισμού. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία μεταξύ όλων σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και ιδίω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε ποια είναι τα θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Πάρα πολλέ φορέ. Πολλά μεγάλα αθλητικά γεγονότα, ιδίω αγώνε ποδοσφαίρου, λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα που έχει το αθλητισμό και τα αθλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι ικανοποιημένο με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τι προτάσει που προήλθαν από τη συζήτηση και συμφωνώ με τον Ιβο Μπέλετ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και να έχουμε κάποιο κεντρικό φορέα που μπορούν να συλλέγονται όλα αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τα προβλήματα διαφθορά και στισήματο. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε χώρα δεν ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στην διπλανή χώρα και αυτή τη στιγμή προσκρούμε και στην αρχή της επικουρικότητας για να αποκτήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Θέλω λοιπόν να πω στην κυρία Επίτροπο ότι την ευχαριστώ για την πρωτοβουλία της και για τη συνεργασία που έχετε προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι μια καλή μέρα για να σταματήσει το σύστημα των αγώνων. Ευχαριστώ, λέει ο Η κυρία Σίνκλερ θέλει να σας ε, κάνει μια ερώτηση με τη διαδικασία της μπλε κάρτας, εάν δεν έχετε αντίρρηση. Κυρία Σίνκλερ, σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφός μου μίλησε για την ακαιρεότητα των αθλητικών αγώνων. Μήπως πρέπει να σκεφτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε σε επίπεδο ακαιρεότητας με την τελευταία της απόφαση, την απόφαση Μπόσμαν, η οποία έχει δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί αυτό έχει πάρει τον πλούτο από πολλές μικρές αθλητικές ενώσεις και τον έχει φέρει στις μεγάλες ομάδες και έχει οδηγήσει σε δύο κατηγορίες ποδοσφαιριστών, καλοπληρωμένων και κακοπληρωμένων. Εκεί είναι που το οργανωμένο έγκλημα στοχεύει τους κακοπληρωμένους ε, ποδοσφαιριστές και στις χαμηλότερες κατηγορίες γίνεται το μεγαλύτερο μέρος της διαφθοράς και όλα αυτά οφείλονται στην απόφαση Μπόσμαν. Ευχαριστώ κύριος Λόκεγκάρτ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόβλημα που ανέφερε η κυρία Σίνκλερ υπάρχει. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί όταν μόνο οι μεγάλες ομάδες έχουν όλα τα χρήματα και οι μικρότερες ομάδες δεν έχουν πόρους, βλέπουμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση και χειραγωγία των αγώνων σε χαμηλότερες κατηγορίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει και σε πιο ψηλά επίπεδα. Δεν μπορείτε να θεωρήσετε ότι οι μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες δεν καλύπτονται. Ο Ιταλός Πρωθυπουργό το είπε πρόσφατα. Όλη λέει η πρώτη λίγα της Ιταλίας θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί για δύο ή τρία χρόνια για να εξαλειφθεί το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Συσσωρεύονται τα χρήματα στις μεγάλες ομάδες και από την άλλη πλευρά έχετε τις ε, χαμηλότερες κατηγορίες όπου είναι ευεπίφοροι σε προσελητισμό από τα συνδικάτα του εγκλήματος οι ποδοσφαιριστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λόκεργαρτ για τους Πρασίνους και την Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Ο κύριος Τεβάρσ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Ήδη εδώ και πολλά χρόνια υπήρξαν ενδείξεις στα κράτη-μέλη για επαναλαμβανόμενα προβλήματα και υπήρξαν και δικαστικές διώξεις ακόμα για, τους, για το γεγονός ότι υπήρξαν στη σήματα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και σε άλλα αθλήματα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε μετά από τις τελευταίες έρευνες της Ευρωπόλ ότι έχει τεράστια έκταση το πρόβλημα αυτό και ότι υπάρχουν και διαμεθοριακά δίκτυα εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε δύο θέματα. Πρώτα, ότι υπάρχει ένα θέμα σύνδεσης με τις ε, οργανώσεις εγκληματικού χαρακτήρα και επομένως εδώ θα πρέπει να έχουμε μια νομική βάση να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης πρόκειται για ένα διαμεθοριακό πρόβλημα το οποίο καλύπτεται αυτή τη στιγμή από την νομοθεσία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι κοινό σε όλους μας μέσα στην κοινωνία μας και ιδίως αυτό αφορά τις αθλητικές ενώσεις και τους αθλητικούς συλλόγους. Πρέπει να συνεργαστούν αυτοί οι σύλλογοι με τις ευρωπαϊκές αρχές για να υπάρξει κάποια εξυγίανση στον αθλητικό τομέα. Δεν μπορούν οι αθλητικοί σύλλογοι που ζητούν την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά για να έχουν ελευθερία σε χρήση και διακίνηση ποδοσφαιριστών να μπορούν να δίνουν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε χώρες όπως είναι η Λευκορωσία που δεν είναι μια χώρα που τηρεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πολλές φορές είναι γνωστό ότι πουλιούνται εκεί τα πρωταθλήματα. Μετά λοιπόν από τις συστάσεις που έχουν γίνει για την πρόληψη της λεύκανης χρήματος και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτά και σε επίπεδο αθλητικών αγώνων. Δεν είναι ένα θέμα φυσικά το οποίο αφορά μοναχά τον αθλητισμό. Θα ήθελα να πω ότι προφανώς είναι πολιτιστικά πάρα πολύ σημαντικός ο αθλητισμός στις ε, κοινωνίες μας και δεν πρέπει να θεωρηθεί μονάχα ως ένας στεγανός χώρος που έχει να κάνει με τα οικονομικά συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε για τους συντηρητικούς δύο λεπτά. Η κυρία Μακκλάρκιν. Αγαπητοί συναδελφοί, καλωσορίζω το ψήφισμα για το στήσιμο των αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό το στήσιμο των αγώνων αποτελεί μία απειλή πανταχού παρούσα στον τομέα του αθλητισμού και η έρευνα της Europol ε, ε, ανακάλυψε ανησυχητικά ε, στοιχεία και πολλοί από εμά έχουμε σοκαριστεί από τα στοιχεία που διαπιστώσαμε. 380, ε, 380 ποδοσφαιρικοί αγώντε θεωρούνται υπόπτη στην Ευρώπη. Αυτό επηρεάζει όχι μόνο τα ανώτερα επίπεδα του αθλητισμού, αλλά σε πολλά επίπεδα ε, έχουμε και στήσιμο αγώνων σε χαμηλότερες κατηγορίες σε όλη την Ευρώπη από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι υπέρ της αυτονομίας του αθλητισμού. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να παρεμβαίνουμε πάρα πολύ στους αθλητικούς συλλόγους, διότι ούτως ή άλλως έχουν από μόνοι τους τρόπο να επιλύουν τα προβλήματά τους. Ωστόσο, αν είναι τόσο ενδημική και διαδεδομένη η διαφθορά όπως διαφαίνεται από τη συγκεκριμένη έρευνα, ε, είναι καθήκον μας να δούμε τι μέτρα πρέπει να λάβουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Αυτοί οι οποίοι ε, κρύβονται πίσω από το στήσιμο των αγώνων είναι συνήθως ε, συνδεδεμένοι με το οργανωμένο έγκλημα. Μπορεί να είναι οργα... οργανώσεις εκτός Ευρώπης ή και εντός Ευρώπης. Είτε εντός όμως είτε εκτός συνόρων βρίσκονται θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει στήσιμο αγώνων στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν είναι ζωτική σημασία να ανταλλάσσονται πληροφορίε ε, για την καταπολέμηση τη διαφθορά και του συστήματο των αγώνων στον αθλητισμό και θα πρέπει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί δεν είναι μόνο εσωτερικό ζήτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ακαιρεότητα είναι επίση πολύ σημαντική και για την βιομηχανία των στοιχημάτων. Ε, πολλές φορές ε, ε, το στήσιμο των αγώνων ε, οδηγεί στη διαφθορά και στο, στα στοιχήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε προκειμένου να προστατεύσουμε την ακυρεότητα του αθλητισμού, τον οποίο αγαπούμε όλοι. Ευχαριστούμε κυρία Μακλάρκιν. Κύριε Μπάτεν, έτοιμος. Σα είδα να έρχεστε τρεχάλα στο διάδρομο. Είστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Έχετε το λόγο. Ε, ε, Τρεχάλα αλλά δεν είναι προπόνηση για το ποδόσφαιρο. Δυστυχώ. Εγώ ευχαρίστω να παραδεχτώ ότι δεν ξέρω τίποτα για τον αθλητισμό, αλλά ξέρω κάποια πράγματα για το στήσιμο αγώνων. Να σας πω πρώτα απ' όλα πω ε, εδώ πέρα απαιτείται μια ειδική μονάδα για την καταπολέμηση του στήσιματο. Εμείς έχουμε ήδη μια ειδική μονάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγεται αστυνομία. Τούτου λεχθέντος βεβαίως Είχα δει και εγώ κάποια στημένα. Το 1975 συγκεκριμένα ήταν ε, στημένο το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ε, ε, είσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μυστικές υπηρεσίες να χρηματοδοτούν ΜΜΕ ήταν λοιπόν στημένο. Στημένο ήταν και το δημοψήφισμα το 1992 στη Δανία, αλλά βγήκε λάθος αποτέλεσμα και τους είπαν ξαναπαίξτε τον αγώνα μέχρι να βγει αυτό που θέμε. Στημένο ήταν και στην Γαλλία και στην Ολλανδία για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, που και εκεί πέρα βγήκε λάθος αποτέλεσμα, αλλά τι έκαναν, άλλαξαν τους κανόνες του παιχνιδιού εκ των υστέρων και λένε «Α, συμφωνήσατε». Και στημένο και στην Ιρλανδία, όταν ε, έβγαλαν και αυτοί λάθος ε, αποτέλεσμα για τη συνθήκη της Λισαβόνας και έπρεπε να ξαναπαίξουν μέχρι να βγει το σωστό αποτέλεσμα. Οπότε αν είναι να ερευνήσουμε τα στημένα, προτείνω να ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε. Ο ε, κύριος Λόκεγκαρντ έχει ένα ερώτημα με την μπλε κάρτα. Το δέχεστε? Ναι. Κύριε Λόκεγκαρντ, έχετε το λόγο. Ο συνάδελφός μου πράγματι απέδειξε πως δεν έχει ιδέα από αθλητισμό. Εξώ και το ερώτημά μου. Εάν φύγουμε από τις πολιτικές πτυχές ε, της ομιλίας σας, αναγνωρίζετε πως ε, εάν είναι κανείς να καταπολεμήσει το διεθνές έγκλημα δεν επαρκεί μια εθνική αστυνομία. Εάν όλες οι άλλες ε, ε, αστυνομίες θέλουν διεθνή συνεργασία, δεν αναγνωρίζετε πώς απαιτείται αυτή. Κύριε Μπάτεν, ναι, ναι, βεβαίως παραδέχομαι πως δεν ξέρω τίποτα για τον αθλητισμό, δεν παριστάνω ότι ξέρω. Αλλά για το διεθνές έγκλημα υπάρχει ήδη ε, ένας αρμόδιος φορέας και λέγεται Ιντερπόλ. Και οι εθνικές μας αστυνομίες διώκουν ε, το έγκλημα μέσα στο κάθε κράτος μέλος. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι γιατί χρειάζεται και ένας νέος φορέας όταν υπάρχουν ήδη αστυνομίες και η Ιντερπολ. Δεν ξέρω γιατί φαντάζεστε πως κάποιος άλλος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πιο αποτελεσματικός από τους υπόλοιπους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Μπάτεν για την Ενωμένη Αριστερά τώρα. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσφάτως η Europol ανακάλυψε ένα ε, οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έστησε πάνω από 380 αγώνες, 425 ε, διαιτητές, αθλητικοί παράγοντες κλπ. αποτελούν αντικείμενο έρευνος και συνελήφθησαν και αρκετοί. Χαιρόμαστε που αρχίζουμε να επενδύουμε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον αθλητισμό. Αλλά το θέμα όμως τι γίνεται με την ε, απελευθέρωση του αθλητισμού και των αθλητικών δραστηριοτήτων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 Ε, δίνουμε όφελο στις καλές προθέσεις αλλά δεν προτείνουμε συγκεκριμένες βιώσιμες λύσεις για τον αθλητισμό. Η φυσική άσκηση είναι πολύ σημαντική για την ε, υγεία του ανθρώπου σε όλα τα στάδια της ζωής του διότι αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα του σεβασμού του άλλου και μαθαίνουμε πώς να ζούμε σε ευγενή άμυλα γι' αυτό και ακριβώς είναι απαραίτητο να φύγουμε από αυτή τη λογική του εμπορίου που θέτει τον έναν ενάντια στον άλλον και ευνοούν αυτές τις μορφές οργανωμένου έγκληματος που έχουν καταλάβει πολύ καλά πώς ε, οι επιχειρήσεις, ε, οι sport business ε, βοηθούν τη συμφέροντά τους. Και επίσης θα πρέπει ε, να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δρούν χωρίς κανένα σεβασμό των κανόνων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θέσουμε τουλάχιστον κάποια ελάχιστα όρια ώστε τα στοιχήματα τουλάχιστον στον αθλητισμό να μην ε, ε, ξεφεύγουν από τα όρια. Θα πρέπει να υπάρχει ε, αυστηρός κανονισμός ε, και πειθαρχία για τους αθλητικούς συλλόγους και να επιβάλλονται αυστηρέ ποινέ ε, για όλους όσους παραβιάζουν τα όρια και να υπάρχει και ευθύνη από πλευρά τραπεζών που υποστηρίζουν ε, αθλητικούς ε, συλλόγους που είναι σχεδόν χρεοκοπημένοι. Και θα πρέπει να μην μείνουμε μόνο στις καλές προθέσεις. Είναι κρίμα, γι' αυτό και εμείς θα απόσχουμε του ψηφίσματο, γιατί είναι κρίμα. Από τους μη εγγεγραμμένους, για 1,5 λεπτό, η κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι αγαπώ τον αθλητισμό, έχω και διαρκεία εισιτήριο και παρακολουθώ όλα τα αθλητικά γεγονότα, ακόμα και μικρούς συλλόγους. Πολλοί αποκαλούν το ποδόσφαιρο το όμορφο, το όμορφο άθλημα, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται το ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει από τα όρια. Από ό,τι φαίνεται πάνω από 10 αθλητικοί αγώνες στην Ευρώπη κάθε εβδομάδα είναι στημένοι. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι εκπληκτικά, αλλά δεν αρκεί να δούμε το θέμα αυτό μόνο από ευρωπαϊκή σκοπιά. Μπορούμε να εμπιστευτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η οποία ε, πρέπει να θέλει να καταπολεμήσει τη διαφθορά για να καταπολεμήσει τα προβλήματα στον αθλητισμό. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και θα πρέπει όλοι να τακτοποιήσουν τα εσωτερικά τους. Αλλιώς πώς περιμένουμε να έχουμε ε, αλλαγές. Στη χώρα μου υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα ε, για ε, τον τρόπο με τον οποίο αγοράζονται οι διάφορες ομάδες και έτσι πολύ καλές ομάδες πέφτουν σε λάθος χέρια. Δυστυχώς ε, δεν υπάρχει κατάλληλη παιδεία και κατάλληλη προστασία και δεν αρκεί μόνο η έρευνα της Europol. Ε, η UEFA έχει πολύ περισσότερες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως η έρευνα μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρκεί. Θα πρέπει οι εθνικές κυβερνήσεις να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα του ποδοσφαίρου δια μιας, διότι εγώ πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει και πάλι ένα όμορφο άθλημα. Να περάσουμε τώρα στους υπόλοιπου ομιλητές. Για δύο λεπτά, ο κύριος Κούρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για τα όσα δήλωσε εδώ στην αίθουσα σήμερα το πρωί και για τα όσα έκανε και σκοπεύει να κάνει στο μέλλον για τον αθλητισμό. Πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερο σημαντικό, αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα. Ο αθλητισμός θεωρείται η ευγενής άμυλα μεταξύ ανθρώπων και λαών. Η αθλητική δραστηριότητα είχε και ιερό χαρακτήρα στην αρχαιότητα και αντίθετα με σήμερα σταματούσαν οι εμπόλεμες ε, ε, σειράξεις και ε, το μετάλλιο ήταν απλώς το βραβείο για τον καλύτερο και όχι για όποιον είχε κοροϊδέψει καλύτερα ή όποιον είχε διαφθείρει τον αντίπαλό του. Σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμό των εθνικών δραστηριοτήτων και των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά επίση γνωρίζουμε ότι το μέτρο αυτό από μόνο του δεν αρκεί και δεν θα αρκέσει ούτε στο μέλλον. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη παιδεία στου νέου πρόληψη, να υπάρχει ε, κατάλληλη εκμάθηση του τι είναι αθλητισμό και να αποτελέσει αυτό την κατάλληλη απάντηση και με τη συμμετοχή των αθλητικών συλλόγων. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζονται μία σειρά από πρωτοβουλίε και σημεία τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε, αλλά θα πρέπει να δράσουμε πολύ γρήγορα, διότι αυξάνεται ο αριθμός νοστιμένων αγώνων. Οι νέοι ε, μεγαλώνουν με μία λανθασμένη αντίληψη για την κοινωνία, διότι ο αθλητισμός βοηθά να κερδίσει ο καλύτερο επιβεβαιώνω και πάλι, και όχι όποιο έχει χρήματα για να στοιχηματίσει καλύτερα. Κυρία Επίτροπε, πρέπει να βιαστούμε πραγματικά, διότι αν διαφθαρεί ακόμα περισσότερο ο θα είναι πολύ πιο δύσκολο να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να εξηγήσουμε στους νέους μας γιατί αξίζει τον κόπο να δεσμευθεί κάτι σε κάτι, σε κάτι σωστό. Κύριε Σκούρια, ο κύριος Βάγκελ θέλει να σας ε, θέσει μια ερώτηση με τη διαδικασία της και μπλε κάρτας. Αγαπητές συνάδελφε Σκούρια, είμαι πίσω σας με χαροποιεί πολύ που μιλήσατε και για την ε, δεοντολογική, την ηθική πλευρά του αθλητισμού και την ανάγκη της δράσης υπέρ των νέων στον ε, τομέα αυτό. Θα ήθελα εδώ να έχω την άποψή σας, γιατί η υπερεμπορευματοποίηση των, ε, του αθλητισμού συνεχίζεται και υπάρχουν τεράστια ποσά τα οποία παίρνουν οι αθλητές και τα οποία υποσκάπτουν κάθε μορφή ε, πειθαρχίας για τους αθλητές. Εμείς έχουμε καταθέσει ψηφίσματα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει η, ένας αποκλισμός του ποδοσφαίρου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες γιατί είναι ένα άθλημα όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα. Μήπως θα πρέπει να θέσουμε κάποια όρια στην εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, Σκούρια. Ναι, συμφωνώ με τον συνάδελφο και για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να μην καταργηθεί η ελεύθερη πάλι που είναι ένα από τα πιο αρχαία αθλήματα τα οποία ε, αναδεικνύουν τον αθλητισμό ε, πέραν της ε, φυσικής επαφής. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο εμπεριβοματοποιείται ο αθλητισμός και ποιος είναι ο στόχος ε, της πραγματικής χορηγίας στον αθλητισμό. Και θεωρώ ότι εδώ είναι ο κατάλληλος χώρος για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε κατάλληλες λύσεις, διότι εδώ ε, Είμαστε 27, πολύ σύντομα και 28 χώρες ε, που έχουμε καθένα καθένας τις διαφορετικές μας εμπειρίες και μπορούμε να έχουμε μια πολύ σημαντική συνεισφορά για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να επιλύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Εντάξει. Δίνω το λόγο για 1,5 λεπτό στην κυρία Μπόσκουρτ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Εγώ ανησυχώ για την κυριότητα του αθλητισμού, για την ασφάλεια των πολιτών μας και ανησυχώ για την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων καθώς το οργανωμένο έγκλημα διεισδύει στον αθλητισμό στην Ευρώπη. Τα σοκαριστικά αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπόλ αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο δίκτυο οργανώσεων που έστησαν εκατοντάδες αγώνες στην Ευρώπη. Το στήσιμο των αγώνων είναι ένα νέο έγκλημα με υψηλή απόδοση, χαμηλό βαθμό ανείχνευσης ε, και χαμηλές ποινές και έτσι μπορούν να ξεπληθούν χρήματα παραδείγματος χάρη από την ε, ε, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών. Γνωρίζουμε λοιπόν το τι συμβαίνει, αλλά θα θέλαμε σήμερα να ακούσουμε από εσά πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος στο θέμα αυτό. Αναφέρατε την Europol, την Eurojust, αλλά χρειάζονται εργαλεία, έναν ορισμό στο ποινικό δίκαιο και καλύτερη ε, συνεργασία, κυρία Επίτροπε. Κάποια κρατημέλη... Συγγνώμη, συγγνώμη, μπορείτε λίγο... Ε, γιατί με ενοχλείτε. Με συγχωρείτε. Κύριε Ένα, σας παρακαλώ. Κάποια κράτη-μέλη εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση άρνησης και είναι πιο ευάλωτα καθώς δεν αντιλαμβάνονται το στήσιμο ως απειλή και έτσι δημιουργούν καταφύγιο για τους εγκληματίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παίξει ένα πιο ισχυρό συντονιστικό ρόλο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το Συμβούλιο της Ευρώπης να τελειώσει με τη σχετική σύμβαση. Το να περιμένουμε μέχρι το τέλος του 2014 δεν σημαίνει πως θα σταματήσουν και οι εγκληματικές οργανώσεις. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα για να προστατεύσει τους πολίτες μας και να διασφαλίσει την ακαιρεότητα του αθλητισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μποσκούρτ. Για ένα λεπτό ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την πρωτοβουλία αυτή που έχει αναπτύξει, η οποία μου φαίνεται πάρα πολύ χρήσιμη και απαραίτητη. Είναι απαραίτητο να δράσουμε από κοινού για τα θέματα αυτά. Σήμερα μας απασχολεί το θέμα το... του αθλητισμού και οι πιο αρνητικές πτυχές που μπορεί να έχει ο αθλητισμός. Θα είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τη διαφθορά στον αθλητισμό, ώστε να είναι ο ανταγωνισμός σε επίπεδο αθλητικό καθαρός και χωρίς στρεβλώσεις, όπως γινόταν και στην αρχαία Ελλάδα. Αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα θέματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις αρνητικές πτυχές του αθλητισμού, αλλά αυτό δεν επαρκεί για να μας δώσει μια συνολική αντιμετώπιση. 90% αυτό που γίνεται στο, στους αθλητικούς στίβους είναι θετικά στοιχεία. Το αθλητισμός είναι απαραίτητος για τη ζωή πολλών ατόμων. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα στοιχεία που είναι παράπλευρες ζημίες του αθλητισμού δεν πρέπει να σπηλώσουν γενικά την εικόνα του αθλητισμού. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, αλλά θα πρέπει να ξαναφέρουμε στο χώρο της ηθικής τον αθλητισμό, να επαναφέρουμε τις Ολυμπιακές αξίες. Και θα πρέπει να επικρατεί η ιδέα ότι μόνο ο καλύτερος πρέπει να κερδίζει. Έχει το λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Χουγουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να αναφέρω ότι ο συνάδελφος κύριος Παπαστάμκος, ο οποίος δίνει μια δύσκολη μάχη και ευχόμαστε να, βγει δυνατός και να γυρίσει κοντά μας είχε δείξει ενδιαφέρον και είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα και θεώρησα σκόπιμο και υποχρέωσή μας να το αναφέρουμε διότι ήταν από τους ανθρώπους που αγωνιούσε για αυτό το φαινόμενο που σήμερα συζητάμε σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζω τα νεότερα στοιχεία της Europol για τα στημένα παιχνίδια. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ακουμπάει μέχρι και ερασιτεχνικά αθλήματα το πρόβλημα και οι αιτίε οφείλονται κατά τη γνώμη μου στο ότι υπάρχει ακραία εμπορευματοποίηση και η καθιέρωση του νόμιμου και του παράνομου στοιχήματος έβαλε, ε, ε, ε, έσκαψε τα θεμέλια ενός, των αθλημάτων και κυρίως του ποδοσφαίρου. Υπάρχει πρόβλημα με τις εθνικές αρχές που είτε δεν θέλουν είτε αδυνατούν να πάρουν μέτρα. Το αυτοδίκητο που επικαλούνται πολλές φορές, κυρία Επίτροπε, δεν πρέπει να αποτελέσει άλοθη για να προχωρήσουμε σε αυστηρά μέτρα, κυρώσεις προκειμένου να υπερασπίσουμε δεν έχω αυταπάτες στο μέτρο του δυνατού και να διατηρήσουμε τον αθλητισμό και τα ιδεώδη του για τη νέα γενιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χουντή. Για 1,5 λεπτό η κυρία Ματιού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να διαλύουμε τα εγκληματικά δίκτυα τα οποία έχουν στήσει 380 αγώνες και πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπόλ για την επιτυχία που είχε στον τομέα αυτό και επίσης ήταν πολύ θετική και η εκπαίδευση των ε, αστυνομικών από την ΕΣΠΟΛ η οποία έχει βοηθήσει πολύ για αυτό το θέμα και η Eurojust έχει κάνει σημαντικό αγώνα για να μπορέσει να εξαρθρώσει τα εγκληματικά αυτά δίκτυα που όπως είπατε κυρία Επίτροπε πολλές φορές στείνουν στοιχήματα και αγώνες. Και φυσικά υπάρχουν και μαφιόζικες οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τέτοια στοιχήματα. Εμείς ε, δεχόμαστε με μεγάλη ικανοποίηση την πρόταση της Κομισιόν για μια οδηγία η οποία καταπολεμά τη λεύκανση των χρημάτων. Ελπίζουμε ότι θα έρθει πολύ σύντομα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεγάλη ικανοποίηση εξάλλου δεχόμαστε την οδηγία για την ε, ε, κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα. Είναι όμως απαραίτητο να επενδύσουμε <clears throat> και στην πρόληψη και να εφαρμόσουμε κανόνες δεοντολογίας στον αθλητικό χώρο και μια πολιτική μηδενικής ανοχής. Υπάρχουν πολλοί γνωστοί αθλητές στην Ευρώπη που είναι πιο γνωστοί από τους μεγάλους συγγραφείς ή τους μεγάλους μουσικούς που έχουν σημαδέψει την ιστορία της Ευρώπης. Για τους νέους αυτοί οι αθλητές είναι το υπόδειγμά τους. Το αθλητισμός συγκινεί τις μάζες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάρα πολλοί ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να αριθμίσουμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Ματιέ. Για ένα λεπτό. Η κυρία Σενάλκοβα. Σενάλκοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόσφατη συνέντευξη τύπου της Europol επιβεβαίωσε το πόσο μικρή είναι η κεραιότητα του ε, ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς στείνονται αγώνες και υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Αλλά οι οικονομικές ζημίες είναι πολύ περισσότερες από τις ηθικές ζημίες. Το αθλητισμό στο το ποδόσφαιρο θα πρέπει να θεωρείται ως ένα ιδεώδες για τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά και εγώ σίγουρα είμαι κατά του στισίματος των αγώνων και του οργανωμένου εγκλήματος και την αντιμετώπιση του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι οι χώρες μεμονωμένα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την ε, δεοντολογική πτυχή του αθλητισμού και θα πρέπει το θέμα αυτό να συμπεριληφθεί και στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και με αθλητικούς συλλόγους. Από ό,τι είδαμε τα περισσότερα ε, μένα μάτς ήταν στην Ασία και εμείς ε, έχουμε ε, υποστεί τι συνέπειε εδώ στην Ευρώπη. Επομένω, το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Γι' αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι συνέπειε ε, και των διαδικτυακών στοιχημάτων στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία Σανάλοβα. Ο κύριο Ιακολίνο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αθλητισμός ε, είναι ένα στοιχείο συμμετοχής και είναι ένα στοιχείο το οποίο διδάσκει αξίες κυρίως στους νέους ο αθλητισμός είναι υγιής και ευγενής άμυλα και θα πρέπει να ανταγωνίζονται με τον αντίπαλο όλοι σε επίσης όρις. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, και το ντόπινγκ το οποίο ε, διαφθείρει και δεν θα πρέπει να υπάρχουν και στημένοι αγώνες στον αθλητισμό. Δυστυχώς ο αθλητισμός πλέον σήμερα είναι απλώς επιχείρηση αξία των αγώνων είναι περίπου 100 δισεκατομμύρια ε, και αυτό το στοιχείο θα έπρεπε να μας ε, κάνει να σκεφτούμε όλους. Η διαφθορά πολλές φορές τροφοδοτείται και από τους ασιατικούς παραδόσεις των παράνομων στοιχημάτων και από την ανακύκλωση βρώμικου χρήματος και αυτό πολύ συχνά βρίσκεται στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται λοιπόν για εγκλήματα τα οποία πολλές φορές είναι διασυνοριακά και γι' αυτό ακριβώς ε, είναι απαραίτητη η δικαστική και αστυνομική συνεργασία, είναι σημαντικός ο ρόλος της Europol, ο ρόλος της Eurojust και θα είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή εισαγγελία η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα εγκλήματα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν και μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει και ρατσιστικός ε, ρατσιστικές συγγνώμη, διακρίσεις μεταξύ των ε, αθλητών, διότι όλα αυτά είναι παθολογίας ενός ε, συστήματος που πάσχει και τον οποίο θα πρέπει να θεραπεύσουμε και να το θεραπεύσουμε το συντομότερο δυνατόν. Εγώ είμαι συγητής ε, για την Επιτροπή ΚΡΙΜ και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές είναι πολλές φορές συνδάλματα για τους νέους μας, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να έχουμε έναν αθλητισμό ο οποίος θα είναι καθαρός από τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστώ. Κυρία Μποσκούρτ, έχετε ζητήσει μπλε κάρτα προς τον κύριο Ιακολίνο. Παρακαλώ, κύριε Ιακολίνο, τη δέχεστε. Η κυρία Μποσκούρτ θα σας θέσει την ερώτηση. Uh, yeah. Ε, ο κύριος Γιακολίνο ανέφερε τα μέλη της Επιτροπής ε, ΚΡΙΜ. Εγώ μάλιστα είχα συντάξει ένα σχετικό έγγραφο γιατί θεωρώ πως το θέμα αυτό δεν είναι απλά αθλητικό αλλά είναι σημαντική περίπτωση που πρέπει να απασχολήσει την επιβολή του νόμου και την δικαιοσύνη. Καθώς λοιπόν έχουμε εδώ πέρα πτυχές ε, ξεπλήματος ε, χρήματος και οργανωμένου εγκλήματος, αναρωτιόμουν πώς θα το εντάξει ο κ. Γιακολίνος στην έκθεση του. Αυτή την απάντηση θα ήθελα. Σας ευχαριστώ κ. Γιακολίνο. Βεβαίω και μπορώ να σας απαντήσω. Να καθησυχάσω τη συνάδελφα Μποσκούρτ οι δραστηριότητε αυτέ που αφορούν του τιμένου αγώνε, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, να υπενθυμίσουμε ότι τα πρώτα στοιχεία αφορούν το baseball πριν από 100 χρόνια. Πρόκειται λοιπόν για ένα φαινόμενο το οποίο έχει μακρά πορεία και επομένω αυτά θα τα συμπεριλάβω στην έκθεσή μου διότι θεωρώ ότι η ακαιρεότητα του αθλητισμού και η ευγενή άμυλα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ω αναπόσπαστο στοιχείο ε, και να αποτελούν κανόνα για τη ζωή των νέων ανθρώπων. Ε, γι' αυτό ολοκληρώνω λέγοντας ότι η δικαστική συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πολύ σημαντική για ένα φαινόμενο το οποίο διαχέεται συνεχώς. Ε, δέχομαι λοιπόν την πρόσκληση της συναδέλφου Μποσκούρ και σας διαβεβαιώ ότι το θέμα αυτό θα επισημανθεί δεόντως ε, στην τελική μου έκθεση αλλά και στην ενδιάμεση έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την ε, νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων. Ευχαριστώ. Για λεπτό, Ρέπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς, ισχύει το ότι το οργανωμένο έγκλημα εμπλέκεται στα στοιχήματα και στο στήσιμο των αγώνων και αυτό καταρακώνει την ε, ηθική δομή του αθλητισμού. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα όμως τα οποία κυκλοφορούν. Υπάρχουν χώρες όπου, παραγωγικά στην Ανατολική Ασία, ζηράνουν εκατομμύρια ευρώ σε στοιχήματα και στέλνουν, λογαριασμού, στέλνουν χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές μέσα από πολυπλοκούς ε, διαδρόμους τραπεζικούς. Δεν μπορεί καμιά χώρα λοιπόν από μόνη της να επιλύσει το πρόβλημα αυτό μόνη της. Και νομίζω το απαραίτητο είναι να υπάρξει μια καλύτερη μορφή ελέγχου που να βασίζεται σε ανταλλαγή δεδομένων και να υπάρξει και μια καλύτερη κάλυψη <clears throat> και εποπτεία των ε, χώρων όπου λαμβάνουν χώρα οι αθλητικοί αγώνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για μισή λεπτό. Ο κύριος Φίσας. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για να αντιμετωπιστεί τον τοπάρισμο, αλλά μονάχα τα τελευταία χρόνια. Τώρα πρέπει να κάνουμε ακριβώ το ίδιο και με το στήσιμο των αγώνων, που είναι μια μάστιγα σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού. Είναι οι παράγοντε, οι διαιτητέ, αλλά και οι παίκτε του ποδοσφαίρου που εμπλέκονται σε, αυτά τα, σε αυτές τις εγκληματικές ενέργειες. Έχουν ήδη προταθεί ορισμένα μέτρα. Να υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα στου οργανωτές των αγώνων ώστε να μπορούν να σταματήσουν τα στοιχήματα που θεωρούν ότι δεν είναι πρέποντα. Επίσης να θεωρείται αδίκημα οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς στον αθλητισμό. Συνεργασία με τρίτες χώρες για τον αγώνα κατά του στισίματος των αποτελεσμάτων και της διαφθοράς στον αθλητισμό. Επίσης να ζητούμε από την Ευρωπόλ να εργάζεται με κοινέ ομάδες και μαζί με την Ευρωσάστ για να ελέγχει και να διερευνά τον, ε, τη διαφθορά στον αθλητισμό. Οι αρχές επίσης θα πρέπει να ελέγχουν όλα, <clears throat> όλες τις συναλλαγές που έχουν να κάνουν με μεταγραφές πολυδοσφαιριστών για να αποτρέπεται η έκπληση χρημάτων. Είναι σημαντική η διακυβέρνηση στον τομέα αυτό. Η διαφθορά γίνεται κυρίως όταν δεν παίρνουν την κατάλληλη αμοιβή οι αθλητές. Επίσης είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ε, παικτών ώστε να μπορούν να κατανοούν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που προχωρούνται από τη διαφθαρά αυτή. Και ζητώ από την Κομισιόν να προχωρήσει σε μια πρόταση βελτίστων πρακτικών για, να, για το επόμενο ήδη έτο πριν από τι ευρωεκλογέ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Παπα-Νικόλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το φαινόμενο της διαφθοράς στον αθλητισμό δεν είναι καινούριο. Ήδη η Ευρώπη απασχολήθηκε για σχετικά θέματα από, τη δεκαετία του 80, θυμίζω το σκάνδαλο το Τονέρο στην Ιταλία και άλλα σε άλλες χώρες, μέχρι και πρόσφατα στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε, ε, έχουμε έρευνα για διαφθορά ε, ίσως σε αγώνα πυγμαχίας. Ε, και βεβαίως η διαφθορά στον αθλητισμό αφορά κυρίως και την Ευρώπη. Αυτό προκύπτει και από τα νούμερα της Europol, το ανέφεραν προηγουμένως και οι συνάδελφοι. 380 από τους 680 ε, στημένους αγώνες ποδοσφαίρου ε, εντόπισε στην Ευρώπη η Europol αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι η συνθήκη της λισαβόνας δίνει πλέον στην ευρώπη μεγαλύτερη δυνατότητα να επέμβει στα θέματα αυτά και γι' αυτό το θέμα και δύο χρόνια πριν το αναφέρω και εγώ όπως και ο κύριος Κοντή προηγουμένως υπήρξε γραπτή δήλωση ε, του κοινοβουλίου μας που εγκρίθηκε για τη διαφθορά στον αθλητισμό ε, του κυρίου παπαστάνκου του συναδέλφου μας. Ε, γνωρίζουμε τις πρωτοβουλίες τη επιτροπής άκουσα με προσοχή προηγουμένως την κυρία επίτροπο και βεβαίω πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και για την πρόληψη. να δώσω ένα παράδειγμα δεν ξέρω κατά πόσο αισθανόμαστε ότι κάνουμε προληπτικά σωστή εποπτεία και έλεγχο στο ηλεκτρονικό στοίχημα. Η λευκή βίβλος για τον αθλητισμό είναι σημαντική. Η διακήρυξη της Λευκοσίας του περασμένου Σεπτεμβρίου για τα στημένα είναι πολύ σημαντική και βεβαίως και η ανακοίνωση δύο χρόνια πριν της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Διάσταση στον Αθλητισμό. Ε, η Ευρώπη είναι περήφανη για τον αθλητισμό της, κύριε Πρόεδρε. Αποτελεί μέρος της ηθικής της και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριο Κούρσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, στον αθλητισμό. Η διαφθορά νομίζω υπονομεύει τις αξίες του αθλητισμού και ο αθλητισμός είναι μία από τις πιο ευχάριστες δραστηριότητες για όλους μας. Και Ακούσαμε βεβαίως πως όλα αυτά είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου και πρέπει να κάνουμε περισσότερα και στην ε, Πολωνία σε έναν βαθμό προσπαθήσαμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο και θα θυμάστε πως είχαμε προβλήματα διαφθοράς ε, κάτι αγώνες με απίθανα σκορ που τελείωναν 7-1 κτλ. Ξέρουμε πως ο Σμπίνιεφ Σμπρόφ, ο πρώην ε, Υπουργό Δικαιοσύνη, ε, έφερε ένα νόμο που αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό, αλλά ε, υπονομεύτηκε η αρχή της αλληλεγγύης. Είδαν πως υπήρχαν προβλήματα διαφθοράς και δωροδοκίων, οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αστυνομιών όλων των χωρών και της κατάσχεσης ε, των ε, προϊόντων του εγκλήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με την διαδικασία και έτσι έχουν ζητήσει κάποιοι τον λόγο. Ο η κυρία Σουντέσχη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές ε, νομικές διατάξεις για διάφορα θέματα και βεβαίω αυτό σημαίνει πως ε, στο θέμα που μας απασχολεί πρέπει να υπάρξει κάποια διαφάνεια. Υπήρχαν στημένοι αγώνες και στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα. Τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί και προφανώς πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να γενικεύουμε, αλλά ξέρουμε πως υπάρχει διαφθορά και έτσι υπονομεύεται η αρχή του εφαγωνίζεστε. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποιε ε, είναι οι λύσεις για να καταπολεμηθεί η διαφθορά στον αθλητισμό και πότε θα μπορέσουμε να δούμε συγκεκριμένε προτάσεις. Σα. ευχαριστώ. Κύριος ε, Μάτσο. Το σκάνδαλο αυτό και τα άλλα στον αθλητισμό επανεμφανίζονται ε, τακτικά. Βεβαίω, 96 σχεδόν θα λέγαμε αφορούν ε, ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ε, υπάρχουν διάφορα μέτρα, το κοινό είναι πιο υποψιασμένο, η εξέλιξη της ε, τεχνολογίας και οι δυνατότητες να στοιχηματίσει κανείς από το διαδίκτυο ευνοούν αυτές τις ε, ε, δυνα... Ε, πιθανότητες να στηθεί ένας αγώνας και βέβαιως πρέπει να καταπολεμήσουμε το στήσιμο των αγώνων και βεβαίως απαιτείται και εκπαίδευση των ε, συμμετεχόντων για να ισχύσει το ευαγωνίζεσθε και η νομοποίηση του σχήματος μπορεί να εμποδίσει ένα μέρος του προβλήματος γιατί μετά δεν θα έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον αυτή η διαφθορά. Μάλιστα. Περνάμε στον επόμενο μελτή. Οι αστυνομίες ε, συνεργάζονται όσον αφορά την ε, καταπολέμηση του στισίματος, αλλά το ίδιο κάνει και το οργανωμένο έγκλημα. υπήρχε μια οργάνωση στην ε, Σιγκαπούρη που ε, έστεινε αγώνες σε 15 χώρες και είχε 700 διαιτητές στην διάθεσή της και στην Ουγγαρία. Το ίδιο μια ουγγρική εγκληματική ομάδα είχε εμπλακεί σε στήσιμο αγώνων μέσω Ανατολικής Ασίας. και στοιχημάτιζαν κάποιοι από 50 έως 100.000 ευρώ και κέρδιζαν τα δεκαπλάσια. Ερευνήθηκε ένας αγώνας μεταξύ Αργεντινής και Βολιβίας το Δεκέμβριο του 2008 και το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε στην ε, ε, παράταση με ένα πέναλτι συγκεκριμένα. Οπότε πρέπει να καταπολεμήσουμε εδώ πέρα τις πρακτικές αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν επιληφθεί αυτού του μεγάλου θέματος. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση σε όλο τον κόσμο ο αθλητισμός και είναι και ένας μεγάλος πειρασμός να κερδίσει κανείς χρήματα με τρόπους οι οποίοι δεν είναι θεμητοί. Οι συνάδελφοί μου έχουν αναφερθεί στο θέμα αυτό, αλλά αυτό δεν αφορά μοναχά το ποδόσφαιρο. Το αθλητισμός είναι κεφαλαιόδου σημασίας για τους νέους. Είναι απαραίτητο να υπάρξει προστασία των νέων αθλητών και είναι ένας τρόπος να δοθεί μέλλον σε άτομα που προερχόνται από μειονακτικά κοινωνικά στρώματα. Στην Ασία γίνονται τα στοιχήματα, αλλά το αποτέλεσμα γίνεται αισθητό στην Ευρώπη. Θα πρέπει να απαγορευτεί όταν είναι νέοι και ανήλικοι οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε αγώνες να γίνονται στοιχήματα και θα πρέπει να υπάρξουν ειδικέ μονάδες που θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σα λέω και πάλι ότι πρέπει να περιοριστείτε σε ένα λεπτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριος Μπίρκη. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε πως ε, Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας της Europol ε, είναι πως ε, έχουμε μπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος, σημαίνει πως θα, έχουμε μια, θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση του θέματος, ε, μια πολιτική μηδενικής ανοχής, να υπάρξει ένας κώδικας συμπεριφοράς, αλλά πρώτα απ' όλα να είναι ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος στο στήσιμο αγώνων. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για να προφυλάξουμε την ακαιρεότητα του αθλητισμού από το οργανωμένο έγκλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Σβέα είναι επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας συγχαίρω για την στάση σας και την ετοιμότητά σας να δείτε αυτό το ζήτημα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μία μορφή διαφθοράς στον αθλητισμό, αλλά δεν είναι η μόνη. Στην ε, Σλοβενία έχουμε ήδη κάποιες ε, δίκες. Είχαμε κάποιες επιτυχίες στην καταπολέμηση του ε, ντόπινγκ. Το ζήτημα είναι το εάν θα το αφήσουμε στα κράτη-μέλη ή θα το λύσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αρχή της επικουρικότητας δεν επαρκεί. Η διαφθορά είναι διασυνοριακή, γι' αυτό πρέπει να το δούμε το θέμα σε διεθνές επίπεδο. Η Europol θα πρέπει να συντονίσει τις ε, διοκτικές αρχές Αυτά είναι σημαντικά βήματα στην καταπολέμηση της διαφοράς, αλλά δεν επαρκούν. Χρειαζόμαστε ε, λοιπόν ευρωπαϊκά μέτρα και νόμους για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λούχαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο βεβαίως... Ε, σωματική δραστηριότητα αλλά και έχει μια πτυχή η οποία διαμορφώνει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Τι κάνουμε λοιπόν όταν απειλείται ακριβώς αυτός ο χαρακτήρας, όταν οι νέοι βλέπουν την τηλεόραση και τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ε, και τα εθνικά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απέναντι σε αυτή τη μάστιγα. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εφιστεί προσπαθειών μαζί με τα κράτη-μέλη για να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία για τη διαφθορά στον αθλητισμό για να καταλήξουμε σε διεθνείς ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες για να σταματήσουν αυτές τις δραστηριότητες και τέλος να συσταθεί μια διεθνής μονάδα για να ελεγχθεί αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο Βασιλείου για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα αξιότιμα μέλη για την ευκαιρία που μου δίνουν να συζητήσουμε σήμερα εδώ με πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία από τις σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός σήμερα, τους στημένους αγώνες. Oh, από ό,τι βλέπω ανησυχούμε όλοι ιδιαιτέρως. Τους τελευταίους μήνες είδαμε εκθέσεις ε, και άρθρα στον τύπο για πάρα πολλά επεισόδια στημένων αγώνων σε όλη την Ευρώπη. Μάθαμε ότι οι στημένοι αγώνες είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο εκτείνεται σε αρκετές υπήρους και πολλές φορές ε, ε, περιλαμβάνει και το δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος αφορά και μεγάλες ομάδες και μικρότερες ομάδες και περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες, ευάλωτους νέους παίκτες, ε, προπονητές, ακόμα και γονείς, αλλά και πάρα πολλούς άλλους. Όπως είπαν πολλοί από εσά, πρόκειται για διεθνές πρόβλημα, το οποίο απαιτεί μια διεθνή λύση. Οι αθλητικές αρχές έκαναν έκκληση για, σε εμά για να τους βοηθήσουμε να προστατεύσουν ε, τους αγώνες τους. Εγώ τους απάντησα και τους είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να δράσει. Δεν είναι εύκολο να καταπολεμήσει κάποιος ένα τόσο σύνθετο ζήτημα όπως είναι το στήσιμο των αγώνων. Ε, συνεργάζομαι στενά με τους συναδέλφους που είναι υπεύθυνοι για τα στοιχήματα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ώστε να υπάρξει μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Έχουμε ε, ξεκινήσει με κάποιες δραστηριότητες πρόληψης που έχουν γίνει από διάφορους ε, φορείς και έχουμε διευκολύνει και το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, οργανώσεις στοιχημάτων, αστυνομικές δυνάμεις, αθλητικά κινήματα, δικαστικό σύστημα. Αλλά το βασικό καθήκον μας είναι να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία ώστε να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση των στημένων αγώνων σε διεθνές επίπεδο. Η χρηστή διακυβέρνηση είναι εξίσου σημαντική και αυτή τη στιγμή Υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που ασχολείται με θέματα χρηστή διακυβέρνηση στου αθλητικού συλλόγου και θα ε, δημοσιεύσουν τι κατευθυντήριε γραμμέ του το 2014. Ε, γίνεται και μια συζήτηση για μια πιθανή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της χειραγώγησης των αθλητικών εκδηλώσεων. Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Συζητούμε επίσης και με την UNESCO για το πώς μπορούμε να θέσουμε το θέμα της καταπολέμησης των στιμένων αγώνων σε πιο υψηλό επίπεδο στο θεματολόγιο για τον αθλητισμό. Μάλιστα, οι στημένοι αγώνε θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην Παγκόσμια Διάσκεψη Υπουργών Αθλητισμού στο Βερολίνο το Μάιο φέτο. Χρειάζομαι τη στήριξή σα σε αυτή τη διαδικασία και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη θετική συνεισφορά που ε, δώσατε σήμερα στη διάρκεια τη συζήτηση. Η καταπολέμηση των στημένων αγώνων είναι ένα δύσκολο έργο και θα τα καταφέρουμε μόνον παρομένουμε ενωμένοι και είμαστε αποφασισμένοι και συνεργαστούμε προ αυτό το σκοπό. Κύριε Πρόεδρε, πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω ότι δεν θα δεχτώ από κανένα να αποκαλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεφθαρμένη. Και θα ήθελα να ρωτήσω το μέλος, ε, τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος ε, ε χρησιμοποίησε αυτή τη διατύπωση, ε, να ζητήσει συγγνώμη, αλλά αποχώρησε από την αίθουσα αμέσως μετά την παρέμβασή της. Ελπίζω εσεί να μην συμμερίζεστε τι παρατηρήσει τη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πίτροπε. Απλώ θα ήθελα να σα ενημερώσω και εσείς και οι υπόλοιποι βουλευτές ότι το, η ψηφοφορία έχει, ότι έχει κλείσει η συζήτηση καταρχήν και η